Good afternoon and thank you. I'm sorry I'm a bit late. The train was a bit late this morning. Over... Λοιπόν, γεια σας. Δεν ξέρω γιατί απουσιάζουν πολλοί Βρετανοί. Ελπίζω να μην αποστασιοποιείται ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο από την υπηρετική Ευρώπη. Συθετήσουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. ανακοινώσει τη Προέδρου. Υπενθυμίζω σε όλου ότι εκπέμπεται στο διαδίκτυο το, η συνεδρίασή μας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το e-meeting. Υπάρχει και η εφημερίδα μα στο newsletter, ενημερωτικό φυλάδι, ενημερωτικό έντυπο. Λοιπόν, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Υποθέτω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος συνεδριάσεως, θεωρούνται τα πρακτικά ως ε, εγκεκριμένα. Πρώτο βασικό σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα, συζητούμε, θα συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες για την πρόταση οδηγίας, για το νομικό πλαίσιο, για τελωνιακές παραβάσεις και κυρώσεις. Η κυρία Κάλλας είναι η συγγήτρια και θα της δώσω το λόγο έκθεση σχετικά λοιπόν αυτήν την οδηγία. Ευχαριστώ. Έχουμε δέκα συμβαστικές ε, τροπολογίες. Οι συμβαστικές αυτές αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες στα ελληνικά θέματα να καταλάβουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν προσπαθούν να παραβιάσουν τους κανόνες, ότι οι περιστάσεις για την παράβαση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι συμβαστικές λοιπόν λαμβάνουν υπόψη ανησυχίες των κρατών μελών όσον αφορά ευελιξία και αναλογικότητα των μέτρων θέλουν υπάρχει περιθώριο να εφαρμόσουν κυρώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα της υποθέσεως. Έχω απομακρυνθεί πολύ την αρχική μου πρόταση για να συμβεβαστώ με άλλες ομάδες. Όπως είχα προτείνει το οικονομικό κατόφλιο για τη διαφοροποίηση μη εγκληματικών, μη ποινικών και ποινικών κυρώσεων που ακολουθείται σε διάφορα κάτι μέλη, σύμφωνα με την ελέγχη του Κοινοβουλίου αυτή η προσέγγιση, έχουμε δύο συμβαστικέ, όπου δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα, για το επίπεδο των κυρώσεων. Είναι το ένα σημείο διαφωνία. Πρότεινα να βγάλουμε το ελάχιστο πάγιο ποσό για μικροπαραβάσεις διότι τα 150 ευρώ μπορεί να θεωρηθούν δυσανάλογα προς την ίδια την παράβαση. Είτε δεν έχουμε ελάχιστο, ή χαμηλό ελάχιστο θα μπορούσε να είναι αποδεκτό για να ρυθμιστεί το θέμα. Όμως, οι ελάχιστε και μέγιστες κυρώσεις σοβαρές παραβάσει είναι πολύ σημαντικέ, πρέπει να παραμείνουν. Δεν έχει νόημα να υπάρχει διαφορά μεταξύ ελαφρών μικρών παραβάσεων και σοβαρών παραβάσεων. Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό κυρώσεω για τι μεγάλε παραβάσει Όσον αφορά τα επίπεδα αυτά καθε γιατί να πάμε από 50% μέχρι 100% των μη καταβληθέντων δασμών. Αυτή είναι η τρέχουσα πρακτική στα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν τα κριτήρια της αποφυγής καταβολής των δασμών. Το 50% είναι αρκετά υψηλό για να δώσει την αναγκαία ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αν δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία θα δημιουργήσουμε πραγματικές διαφορές για τις επιχειρήσεις στην ενία αγορά Ελπίζω λοιπόν να το λύσουμε αυτό το θέμα και να ψηφίσουμε επιτυχώς την Επιτροπή δοθήσει στις προσπαθίες που καταβάλαμε και των συμβιβασμών που υπευλήθησαν και όλων των προσπαθειών που έγιναν γενικά για αυτό το θέμα. λοιπόν, λέει η Πρόεδρος. Αντώνιο ή Ρομπέρτα. Η Ρομπέρτα Ματσόλα. Α. Όχι. Ρομπέρτα Ματσόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ την Κάγια. Έξοχη δουλειά που έκανε. Βελτίωσε την πρόταση. Συμπεριέλαβε τα περισσότερα σχόλια των σκιωδών. Δεν αποτελεί μυστικό ότι πολλοί από εμά, όπω και η ομάδα μου, είχαμε ισχυρότατε επιφυλάξει όσον αφορά την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτιμούμε τα μάλα τι καταβληθήσει προσπάθειε για τι αναγκαίε αλλαγέ για διακομματική συμφωνία. Επίσης είναι πασίγνωστο ότι έχουμε ανησυχίες που εκκρεμούν σχετίζονται με την αρχή της επικουρικότητας οι περισσότερες ανησυχίες. Θα θέλαμε τα κράτη-μέλη και αρμόδιες αρχές αυτών να έχουν την αναγκαία ευκαμψία, ταυτόχρονα όμως να εξασφαλίζουμε ότι η πρόταση θα ευθυγραμμίζει το καθεστώς των κυρώσεων που επιβάλλονται στις τελωνιακές παραβάσεις. Υπό το φως αυτού πρέπει να αρθεί η ελάχιστη κύρωση για μικρο παραβιάσεις του άρθρου 11 και όσον αφορά τις κυρώσεις που σχετίζονται με τα τέλη που δεν έχουν καταβληθεί. Με τους δασμούς που δεν έχουν καταβληθεί. Αυτή η αλλαγή πάει μεγάλη διαφορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για ιδιώτες που διαπράττουν μικρο Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα μου, διότι οι αρμόδιε αρχέ των κρατών μέλων πιστεύουμε μπορούν να αποφασίσουν για παραβιάσει των τελωνιακών δασμών και την επιβολή των αναγκαίων κυρώσεων, κατά περίπτωση. Γι' αυτό εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αναγκαία ευελιξία, τόσο ώστε αυτέ οι αρχέ να μπορούν να κάνουν τη δουλειά του σωστά. Τώρα, σε αυτό το στάδιο που είμαστε τη νομοθετική διαδικασία, δεν θέλουμε να εκφράσουμε ευχολόγιο για τα αποτελέσματα τη προτάσεως κατανοούμε ότι υπάρχει ένα κείμενο για τελικό συμβιβασμό που είναι σχεδόν έτοιμο και αντικατοπτρίζονται κάποιε ανησυχίε τη ομάδα. Όμω θα έπρεπε να έχουμε σαν στόχο να ρυθμίσουμε τι λεπτομέρειε του κειμένου με μικροαλλαγέ, ούτω ώστε η πρόταση αυτή να προωθηθεί δεόντω. Και θα εξαρτάται όταν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να δράσουν. Ω αρμόζει. Η ομάδα μα θα περιμένει το τελικό συμβαστικό κείμενο και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειε ούτω ώστε εμπεριστατωμένα να αποφασίσουμε για την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα στην Επιτροπή. Είμαστε σε συνεχείς επαφές με την εισηγήτρια και θα συνεχιστούν οι επαφές, διότι συνεργαζόμαστε άριστα και ευχαριστούμε και εκείνοι και τους συναδέλφους για την προθυμία επιτεύξεως συνενέσεως ή τουλάχιστον απόψεως που θα συγκεντρώνει την πλειοψηφία σε αυτή την Επιτροπή. Αυτά και ευχαριστώ. Ποιος μιλάει στους ελιστέ τώρα δεν είναι εδώ. Πάμε λοιπόν στον Ντάν Ντάλτον. Ευχαριστώ. Βίκυ, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα. Πάντα δεν δεχτήκαμε τη βάση της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είδαμε να υπάρχουν στοιχεία επιλογής του καταλήλου του πιο βολικού καθεστώτος. Αλλά εμείς ανησυχούμε για την επικουρικότητα του του λεχθέντος. Κάποιες από τις προτάσεις του ΕΛΚ για ελάχιστο κατόφλιο κυρώσεων, η πρόταση για μηδέν παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αναλύουμε την πρόταση. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το στηρίξουμε. Γιατί ανησυχώ από αυτού. Δεχόμαστε την υπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποφασίσει εν πρώτης το κατόφλιο. Μπορεί να είναι μηδενικό σήμερα το κατόφλιο στο μέλλον, μπορεί και να μην είναι μηδέν. Άρα ανησυχούμε. Γι' αυτό ακριβώς. Επίσης ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί το λέω αυτό. Διότι σε ένα ψηφιακό κόσμο μιλάμε για ψηφιακή ενιαία αγορά. Πάντα γι' αυτό μιλάμε. Και σε έναν ψηφιακό κόσμο αγοράζει ο κόσμο στο διαδίκτυο πράγματα από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και όταν αγοράζει από χώρα εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω, από τη ΣΥΠΑ, Φερρυπίν, και είναι πάνω από 200 ευρώ αξία του, σου χτυπάει την πόρτα το τελωνίο. Και σου βάζει και πρόστιμο ο τελωνιακό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κάποιες από τις προτάσεις των σοσιαλιστών, δηλαδή ότι το ελάχιστη, η ελάχιστη κύρωση πρέπει να είναι 7.500 ευρώ όταν έχεις ε, παραγγείλει ένα σοτσάκι από τη ΣΥΠΑ, είναι παράξενο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι κάνουμε. Αν στην απίθανη περίπτωση βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί κανείς να μπλέξει φέρνοντας ένα μήλο του Ηνωμένου Βασίλειου στο Βέλγιο. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα τα των τελωνίων να είναι σωστά ρυθμισμένα. Δεν είδα κανένα στοιχείο ότι μας χρειάζεται αυτή η πρόταση. Είναι πρώτης. Αλλά, τούτου λεχθέντος, εξετάζουμε την πρόταση του ΕΛΚ όσον αφορά τι ελάχιστε κυρώσει. Θέλουμε να δούμε, βλέπετε, κατά πόσο μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Όπω είπα, όμω, εξακολουθώ να, μην καταλαβαίνω το αρχικό επιχείρημα, τη βάση, την προσέγγιση δηλαδή. Την υπόθεση τη οποία βασίζεται. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τα 200, τα σορτσάκια που θα αγοράσει με τα 200 ευρώ. Λοιπόν, κάποιο από την ΚΟΕ θέλει να μιλήσει. Όχι. Κάποιος από τους πράσινους μήπως. Αντρές Σουάπ. Αντρές Σουάπ. Όχι από τους πράσινους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω δύο σημεία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την απόφαση του δικαστηρίου του ΠΟΕ δεν μπορούσε παρά να υποβάλει πρόταση ώστε διακόπτεται ο μιλητής χωρίς μικρόφωνο. Κάτι πολύ περίεργο γίνεται με τη διερμηνία. Στο 2 δεν είναι αγγλικά αυτά που ακούγονται. Πολωνικά ήτανε. Sorry, Andreas. Don't worry, don't worry. Συγγνώμη κύριε Σβάμπ. Δεν θα υποστείτε κυρώσεις. Μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. It's coming in my ear, not English. That's, yes, that's better. Thank you. Ναι, καλύτερα τώρα. Ευχαριστώ. Dress. Να ξαναπροσπαθήσετε κύριε Σβάμπ. Από το ΕΛΚ ο κύριος Σβάμπ, όχι τον πράσινο του ΕΛΚ. Λοιπόν και πάλι ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά του, διαιτητη, της απόφασης ε, του σώματος του ΠΟΕ δεν μπορούσε παρά να προσαρμόσει το τελωνιακό δίκαιο όσον αφορά τις κυρώσεις και τα πρόστιμα. Ήταν σαφές ότι τα κράτη-μέλη με πολύ μικρή ικανοποίηση θα δεχόντουσαν μια τέτοια πρόταση και γι' αυτό τρίτον κάπως εκπλήσει το πώς η πρόταση από την Επιτροπή έγινε τελικά. Πιστεύω ότι η συγγήτρια πραγματικά έκανε μεγάλη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Ένα συμβιβασμό όμως που λόγω της κατάστασης της ίδιας κατεπηγόντως ε, έτσι όπως ε, προδιαγράφεται και θα έλεγα ότι ο Επίτροπος είχε έρθει στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή Πρόεδρε και μίλησε για μια στρατηγική για το τελωνιακό δίκαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ για μένα και για την ομάδα μου θα έπρεπε να πω ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε τι έγκυται αυτή η στρατηγική και ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα. Διότι στο τέλος τέλος για τα τελωνιακά θέματα, το τελωνιακό, τελωνιακό δίκαιο είναι αρμόδια τα κράτη-μέλη και πρέπει υποχρεωτικά από πλευρά της Επιτροπής να ληφθεί υπόψη η αποδοχή των προτάσεων από τα κράτη-μέλη και εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μια και οι συμβιβασμοί που έγιναν με αυτή την πρόταση μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. So I I heard... Λοιπόν, νομίζω ότι κάποιος είχε ζητήσει, κάποιος συντονιστής του ΕΛΚ, ζήτησε να καλέσουμε τον αρμόδιο επίτροπο για τα τελωνιακά να επιστρέψει στην Επιτροπή μας να συζητήσει τα τελωνιακά θέματα. Δοθέντων των προβλημάτων που έχουμε με τον τελωνιακό κώδικα της Ένωσης και την κατεξουσιοδότηση πράξη θα ήταν λογικό αυτό. Θα κάνουμε τα δέοντα με τους συντονιστές λοιπόν να το προωθήσουμε αυτό. Άλλος που θέλει να μιλήσει. Κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θέλει να τοποθετηθεί. Α, ορίστε. Λοιπόν, η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σημειώνουμε με θικανοποίησους και ενδιαφέροντος ότι καταλήγεται σε κάποια θέση όσον αφορά το δύσκολο αυτό θέμα. Το παραδεχόμαστε, είναι δυσχερέστατο χαρτοφυλάκιο. Σημείωσα τα αναφερθέντα και αυτό που είπατε ότι θα συζητήσετε με τους συντονιστές για να προσκληθεί ενδεχομένω ο αρμόδιος επίτροπος να έρθει στην επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Και έχουμε συνεχείς ερωτήσεις που καταφθάνουν από τους ενδιαφερομένους για θέματα που αφορούν τον τελωνιακό κώδικα. Δεν μπορεί κανείς να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να το φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το οποίο μας κάνει, μας μπερδεύει. Παλιά μπορούσαμε να το κάνουμε επί σειρά ετών και τώρα έχουμε μπερδευτεί. Λάθος η προσέγγιση. Κακώ είναι ρυθμισμένες σε διάφορες λεπτομέρειες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Η κυρία Κάλλας έχει το λόγο. δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Ξέρω πού βρισκόμαστε συνεργαζόμαστε για να λύσουμε τα θέματα των δύο συμβαστικών, θα καταλήξουμε σε τελική πρόταση εν ευθέτω χρόνο. Καλώ, α προχωρήσουμε. Πάμε στο επόμενο σημείο. Θα συζητήσουμε συμβιβαστικέ τροπολογίες και τροπολογίες για την γνωμοδότηση, για την εντολή, για τριμερή διάλογο, για τον προπολογισμό του 2017. Θα το ψηφίσουμε αυτό αύριο. 19 τροπολογίε υπευλήθησαν και τέσσερις συμβιβαστικέ τροπολογίε είναι αντικείμενο σύμφωνε. Η κυρία Τσάρη έχει το λόγο. κονσάρι. Σα ευχαριστώ πολύ, Προέδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδη για τη συνεργασία τους. Ήταν έκτακτη η συνεργασία μα. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, πράγματι έχουμε 19 τροπολογίε. και δημιουργήσαμε, συντάξαμε πέντε συμβαστικές τροπολογίες τελικά. Τα αποτελέσματα είναι καλά ισορροπημένα πιστεύω. Και διαπιστώσαμε ότι όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, ότι υπάρχει υποστήριξη για την κυκλική οικονομία. Θα πρέπει επίσης να δούμε ότι η προστασία του καταναλωτού θα πρέπει να διευθετηθεί καταλήλως. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν και κυρίως οι διατάξεις για την προστασία του καταναλωτού ε, πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Υπήρχε σύμπνοια όσον αφορά το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι που υπογραμμίζεται. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την αραστή συνεργασία. Ευχαριστώ. Αντώνιο Λόπες Εστουέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για Κονσάρι Κύριε Γιακονσάρη. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για τη στάση, ενεργητική στάση όσον αφορά την αναζήτηση συνενετικών λύσεων. Νομίζω ότι μπορούμε αύριο να έχουμε ένα κείμενο σε σχέση με την ψηφοφορία ισορροπημένο για αυτή τη γνωμοδότηση ως μήνυμα προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών για την πολιτική μας, για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά και τα κονδύλια του 2017 στο αρχικό κείμενο συγχαρητήρια για τη δουλειά και για τις τροπολογίες που δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για μένα, για το ΕΛΚ, ήταν σημαντικό να διατηρήσουμε το πνεύμα της παραγράφου 2 όμως διαγράφοντας θέματα ανταγωνισμού όσον αφορά τα, τις μελλοντικές συμφωνίες, διεθνείς συμφωνίες. Δίνω απόλυτη συμφωνία, σύμφωνη γνώμη για την τροπολογία 1 σε αυτό το θέμα. Άλλα θέματα που μπορούν να υπογραμμιστούν είναι τα δίκτυα για τους καταναλωτές, ευρωπαϊκά δίκτυα για τους καταναλωτές και για το φόρουμ για την ενιαία εσωτερική αγορά στην αντίστοιχη παράγραφο της γνωμοδότησης. Να μην ξεχνάμε ότι οι αρμοδιότητές μας συμπεριλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την αναφορά στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία στην παράγραφο 2 ευθυγραμμιζόμενη με, την, ε, ε, με τα όσα εγκρίθηκαν το 2015 για την κυκλική οικονομία είναι ένα θέμα που κερδίζει η επικαιρότητα κάθε μέρα και ως Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση σε αυτή την πολιτική. Θέλω να συγχαρώ για τις ιδέες που συνεισφέρατε σε αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ. Dalton. ευχαριστώ, Βίκη. Εμείς δεν υποβάλαμε τροπολογίες. Ελπίζαμε η συγγήτρια να λάβει υπόψη τις προτάσεις μας, να κατήσουμε δηλαδή τα ανώτατα όρια. Σε αυτό το στάδιο δυστυχώς αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Άρα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη θέση αυτή. Έχουμε πρόβλημα τη διαδικασία όσον αφορά τις εκθέσεις περί προϋπολογισμού. Εμείς δεν είμαστε κατά σωστή χρηματοδότηση για τα θέματα τη ενιαία αγορά. Το υποστηρίζουμε αυτό, όταν αξίζει τον κόπο να δαπανίσουμε χρήματα. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι κάθε επιτροπή απλώ ετοιμάζει ευχολόγιο συμπληρωματικών δαπανών. Και ουσιαστικά τελικά δημιουργεί το παλιό πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δαπανούμε όλο και περισσότερο χρήματα και δεν εστιαζόμαστε επί των αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά τη διαδικασία. Εάν αυτό δεν αναγνωριστεί, παρόλο που θέλουμε και άλλα χρήματα για την εσωτερική αγορά, αυτό πρέπει να επιτευχθεί με μείωση από άλλους τομείς που ίσως να μην αξίζουν τόσο πολύ χρηματοδότηση. Χωρίς αυτή την προσέγγιση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αλλιώς ξαναμπλέκουμε. Μπαίνουμε στο παλιό παιχνίδι να ζητάμε περισσότερα χρήματα και θα τα πληρώσει τελικά ο φορολογούμενος. Και δεν νομίζω ότι είναι δίκιο. Λοιπόν, δυστυχώς παρόλο που η έκθεση δεν είναι και πολύ κακή, επειδή δεν συμπεριλαμβάνει όμω αυτό, δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να την υποστηρίξουμε. Ο Ντίτερ δεν είναι εδώ. Από την Άλτερ. Άλλος θέλει να μιλήσει για την ΚΟΥΕ, τους πρασίνους, υπάρχει κάποιος με σχόλια και μετά μπορούμε να επιστρέψουμε. Η κυρία Γιακονσάρη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη την πρόταση αυτή. Καταρχήν δεν υπήρχε τροποποίηση, δεν υπήρχε πρόταση τροπολογίας και για να συμπεριληφθεί αυτό το θέμα στις συζητήσεις. Και στη συνέχεια χρειάζεται να γίνει λόγος με πολύ πιο εξειδικευμένο τρόπο για αυτή τη μορφή του προϋπολογισμού που πρέπει να έχει αρκετή ελαστικότητα ώστε να μην χρειάζεται να ρίχνουμε κονδύλια στον προϋπολογισμό αλλά να επικεντρωνόμαστε στο έργο με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν υπήρξε όμως κάποια τροπολογία. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο το πρωί. Ωραία. Ας προχωρήσουμε. Πάμε και γρήγορα μάλιστα. Ο κύριος Ζούλο είναι εδώ. Πριν ξεκινήσουμε Μάρκο, ας περιμένουμε ένα πεντάλεπτο. Ε. Μήπως καταφτάσουν και άλλοι σκιώδεις. Ο Νίκολας είναι εδώ. Η Εύα. Εσείς η Εύα. Και εσείς η Έμα. Ωραία, όλοι εδώ. Ο Μάρκο Ζούλο λοιπόν είναι εισηγητή γνωμοδότη για συνοριακή φορητότητα περιεχομένου του διαδικτύου και των σχετικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Να το μεταφράσω για όσου μα ακούνε, να μπορεί να πάρει το ψηφιακό σου περιεχόμενο μαζί σου όταν ταξιδεύει στην Ευρώπη. Μάρκο, εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησή του. Σου, μάλλον. Θα έχει την καλοσύνη να μα παρουσιάσει λοιπόν το θέμα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Presidente. Ευχαριστώ. Ο κανονισμό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εγγυηθούμε τη φορητότητα του ψηφιακού περιεχομένου σε όλη την Ένωση είναι κάτι σύντομο και σαφέ, με συγκεκριμένου στόχου. Το draft που δόθηκε λοιπόν, χάρη στι συζητήσει των εβδομάδων, περιορίζεται σε κάποια σημεία που θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν περιττέρω. Πάνω απ' όλα πιστεύω ότι η ύπαρξη πληρωμής σε χρήματα σε ρευστό είναι προπόθεση του ώστε ο πάροχο να έχει την υποχρέωση να εγγυάται τελικά τη φορητότητα και θα έχει μια υποχρέωση να εξακριβώνει το κάτω μέλο τη διαμονή ε, του ε, συνδρομητή που είναι προϋπόθεση βασική για να αποφευθεί η κατάχρηση όσον αφορά τον τομέα. Λοιπόν, οι πάροχοι των δωρεάν ε, μάλλον υπηρεσιών θα πρέπει να εξαιρούνται, διότι χωρί σύμβαση ο πάροχο δεν έχει σίγουρα στοιχεία και επαρκή στοιχεία για να εντοπίσει το κάτος μέλο διαμονή του χρήστη. Λοιπόν, λάβαμε υπόψη ότι στην κατάρρευση των φραγμών που εμποδίζουν του Ευρωπαίου πολίτε να μπορούν να απολαύσουν αγαθά και υπηρεσίε που ήδη έχουν αποκτηθεί, είναι απαραίτητο να έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα που ενδεχομένω να είναι αντίθετα. Σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένη θα είναι καλό να λάβουμε υπόψη την προστασία του δικαίματο του δημιουργού και τη λειτουργία των μηχανισμών οικονομικής βιωσιμότητας της οπτικοκουστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη που επιτρέπει μέχρι τώρα ποικιλομορφία πολιτισμική που θα πρέπει να προστατευθεί προς όφελος των ιδίων των πολιτών. Πιστεύω γι' αυτό ότι η φορητότητα σε δυσυνορικό επίπεδο θα πρέπει να μεταμορφωθεί σε μια πανευρωπαϊκή άδεια. Λοιπόν, Λοιπόν, λέει τρία χρόνια από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση. Θα πρέπει να δούμε ότι δεν δημιουργούνται επικίνδυνε ανισορροπίε οικονομικέ όσον αφορά του κατόχου των δικαιωμάτων, των παρόχων των υπηρεσιών και των χρηστών ή υπερβολικό κόστο για οδήποτε συμμετέχον μέλο. Στον κανονισμό θα πρέπει να καθορίσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια την έννοια του κράτου μέλου τη διαμονή, για να μην αφήσουμε περιθώρια αβεβαιότητα ρυθμιστική που θα μπορούσε να δημιουργήσει καταχρήσει όσον αφορά την εφαρμογή των φόρων διατάξεων. Έναντι των πολλών ορισμών τη συνήθου διαμονή, πιστεύω είναι σκόπιμο ο κανονισμό να προβλέπει τα διάφορα επαρκή κριτήρια που θα πρέπει να προβλέπονται για να καθορίσουμε τη διαμονή που να είναι κάτι αναφυσβήτητο για να εφαρμοστεί η αρχή τη ε, φορητότητα. Για να εγγυηθούμε τη μέγιστα λειτουργικότητα λοιπόν του συστήματο, θα πρέπει πρέπει να επιφορτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει τον κατάλογο των κριτηρίων μέσω μια καθιστοδότη πράξη που μπορεί να έχουμε τι κατάλληλε διαβουλεύσει και με του εκπροσώπου των καταναλωτών και με του εκπροσώπου του κόσμου τη βιομηχανία. Λοιπόν, ο καθορισμό του κράτου μέλου τη διαμονή θα πρέπει να γίνεται με αδιαφεσβήτητο τόπο και να μην μπορεί να έχει κάποιο διαμονή σε πάνω από ένα κάτω μέρο να ισχυριστεί τη διαμονή. Η επαλήθευση τη χώρα διαμονή θα πρέπει να γίνει τη στιγμή τη συνδρομή στην υπηρεσία, αλλά και κατόπιν. Με συνεχή τρόπο, αλλά όχι σταθερό. Να μην έχουμε πολύ δυσδυτικό έλεγχο όσον αφορά τον ίδιο το χρήστη. Λοιπόν, ο χρόνο διαρκέ φορητότητα δεν θα πρέπει να περιορίσει συγκεκριμένο αριθμό ημερών, για να μην είναι επιζήμιο για τι κατηγορίε των πολιτών, του οποίου θέλει να προστατεύσει οδηγία. Δηλαδή εκείνους που πηγαίνουν διακοπές για δουλειά, που ταξιδεύουν όπως είναι οι παραμεθόροι εργαζόμενοι και για σπουδές, όπως ε, οι φοιτητές ε, του Έρασμους. Τέλος, οι πάροχοι περιεχομένου που κάνουν δίνουν ε, υπηρεσίες χωρίς χρήματα από, το συνδρομητή θα πρέπει να μπορούν να μπουν στον κανονισμό, να καλυφθούν. Όμω θα πρέπει να συμμορφωθούν με όλε τι διατάξει του κανονισμού για να γίνει αυτό. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα αυτά που απαιτούνται για ε, επαλήθευση τη χώρα διαμονή. Σε αυτή την περίπτωση, για να αποφύγουμε καταχρήση οικονομικέ ζημίε στου δικαιούχου ε, των ε, πνευματικών δικαιωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου. Τώρα, θα πρέπει λοιπόν να γίνει διαμόρφωση των συμβάσεων ε, που γίνονται στον αφορά του παρόχου ε, υπηρεσιών online και χρειάζονται συστήματα αποτελεσματικά επαλήθευση τη συνήθου διαμονή. Θα πρέπει να επεκταθεί από 6, κατά 6-12 μήνε ο χρόνο που προβλέπεται τη θέση ισχύ του παρόντο ε, κανονισμού. Αυτέ είναι οι γενικέ τροποποίησει που έκανα εγώ στην έκθεση και με τα χαρά να ακούσω όλου του κοιόδη και του συναδέλφου που θέλουν να μιλήσουν, γιατί πιστεύω ότι είναι μια έκθεση αρκετά πλήρης και μια καλή ομαδική δουλειά θα επιτρέψει να προτείνουμε στην Επιτροπή την Νομική ένα πάρα πολύ ε, εμπεριστατωμένο κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ρομπέρτα θα μιλήσει εκ μέρους της. Ευχαριστώ πολύ, Βίκη. Όπως πολύ σωστά είπες, ε, είμαι εδώ και αντικαθιστώ την Εύα Πάνοβο, που είναι σκιώδη συγγητρία για αυτό το θέμα. Η Εύα θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή, είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα έχουμε σωστά εργαλεία, τα οποία θα επιτύχουν το θέμα της φορητότητας στην κοινή αγορά. Ε, κανείς δεν χρειάζεται να μας πείσει ότι πρέπει να ισχύει η φορητότητα. Το κείμενο διευκρινίζει ότι η καταβολή υποχρεωτικής εισφοράς σε κάποια κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμβόλαιο ε, με αυτή την έννοια του κειμένου. Ε, ένα άλλο θέμα είναι ότι το να αποφεύγουμε τον έλεγχο δεν βοηθάει. Επίσης, το ίδιο πρόβλημα θα πρέπει να ισχύει και όσους ε, προσφέρουν τις υπηρεσίες, αλλά ε, αυτό θα μπορεί να γίνεται και χωρίς καταβολή φοράς Πάντως, εάν τελικά ασκεί κανείς αυτά τα δικαιώματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να επαληθεύσει, οι συνέπειες θα πρέπει να είναι ίδιες όπως εκείνων των παρόχων που προσφέρουν υπηρεσίες. Ε, επιπλέον, στην τροπολογία υπαριθμών 14 είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι το opt-in είναι ε, μια πρόταση είτε ναι είτε τίποτα. Και πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ο πάροχος δεν μπορεί να επιλέγει εφαρμογές από άλλες περιπτώσεις. Ε, το σημαντικότερο σημείο στον κανονισμό είναι η διαδικασία επαλήθευση, η οποία θα πρέπει να είναι εύκολη τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον πάροχο. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να είναι εύκολο καταναητό που λειτουργεί έχοντας ε, κατά νου ότι οι τεχνολογίες ε, σε πολλές περιπτώσεις αρκούν για την ε, επαλήθευση του τόπου διαμονής. Εμείς θα θέλαμε να βρούμε μια συμβαστική πρόταση ανάμεσα στους 6 και τους 12 μήνες. Η Εύα θέλει να ευχαριστήσει όλους και προσβλέπει στη συνεργασία με τον εισηγητή και με όλους τους άλλους αντέλφους για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και τον ευχαριστώ Τζούλο το συνάδελφο Τζούλο για την ε, ε, έκθεσή του. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία με τη φορητότητα. Εμείς ε, στη φάση συζήτησης, αρχική συζήτηση, έχουμε ήδη εκφράσει την πλήρη υποστήριξή μας στην πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία πρωτοβουλία θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές σε μεγαλύτερες δυνατότητες να χρησιμοποιούν τη φορητότητα και στο εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο του κανονισμού και το Συμβούλιο έχει διεργαστεί από αυτού τους προηγούμενους μήνες για να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τη φορητότητα αποφεύγοντας τις ε, καταχρήσεις και παράλληλα να προστατεύεται και η ιδιωτικότητα των ε, καταναλωτών. Άρα δηλαδή πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαιότητα να ξεπεράσει κανείς τα όρια που τώρα είναι ξεπερασμένα και από την άλλη, από την άλλη να μην διευκολύνουμε τις ε, καταχρήσεις. Να μην υπάρχει δηλαδή ε, δυνατότητα κατάχρησης, να μην μπορούν να το κάνουν κάποιοι όσον αφορά την επικοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικότερο θέμα επί του οποίου πρέπει να εργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες και το Συμβούλιο έχει κάνει από αυτού πολύ καλή δουλειά είναι ο σαφής ορισμός της ε, συνήθους, ε, του συνήθους κανονικού τόπου διαμονής. Ε, αν λυθεί αυτό το θέμα τότε η νομική βάση ε, για τον κανονισμό, θα είναι ισχύουσα, θα είναι αποτελεσματική ε, και θα προστατεύει τα δικαιώματα στα διάφορα κράτη-μέλη. Όσον αφορά στα κριτήρια επαλήθευσης, νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και εκ μέρου του Συμβουλίου και πρέπει να έχουμε κριτήρια τα οποία εύκολα εντοπίζονται, είναι εφαρμόσιμα και παράλληλα ε, προσφέρουν και τη μέγιστη ε, σιγουριά ε, σχετικά με τέτοιου είδους συνδρομές. Η δουλειά του Συμβουλίου είναι πάρα πολύ καλή και πλέον εναπόκειται σε εμά να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όλο αυτό το θέμα. Γιατί από τη στιγμή που έχει ξεκαθαριστεί ε, ποιος, έχει ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο τόπος διαμονής θα προκύψουν ε, άλλες ανησυχίες ε, σχετικά με το χρόνο, τον περιορισμένο χρόνο και με τη δυνατότητα που δίνει σε κάποιον που ζει στο εξωτερικό για κάποιες ε, ημέρες. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Και όπως ακριβώς ε, εντοπίζει κανείς ε, πού ακριβώς βρίσκονται, υπάρχει ο κίνδυνος της ε, παραπίεσης της ιδρυτικότητας των ανθρώπων. Άρα δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά όσον αφορά τον τόπο διαμονής. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που κατά την παραπιεσης της ιδιωτικότητας μου πρέπει να εμβαθύνουμε. Είναι ακριβώς το ότι θα πρέπει να έχουμε κατεξοδότηση πράξης οι οποίες θα μπορούν στην ε, Κομισιό να προσφέρουν τα κριτήρια με τα οποία εντοπίζει κανείς ε, τον ε, τόπο διαμονής. Πρέπει να υπάρχει ένας σαφής κατάλογος όσον αφορά στον κανονισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα επί το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας τις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα δεν έχω σαφή απάντηση παρότι φαίνεται ότι είναι καλύτερο ε, ευθύς εξ αρχής να θέσουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία. Και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο αφορά στους ε, παρόχους ε, δωρεάν περιεχομένου. Το opting in είναι σημαντικό, πρέπει να διατηρηθεί, να ισχύουν τα ίδια κριτήρια με εκείνους που πληρώνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σκόπιμο να προσφέρεται αυτή η δυνατότητα σε πάρα πολλούς ε, ε, δωρεάν, ε, σε παρόχους δωρεάν υπηρεσιών να μπορεί κανείς να ικανοποιήσει τους πελάτες του και στο εξωτερικό και πάντα σεβόμενος κανείς τα κριτήρια που ισχύουν για εκείνους που ε, προσφέρουν περιεχόμενο ε, με κάποια πληρωμή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να περάσουμε στην έγκριση αυτού του κανονισμού. Νομίζω ότι τους προηγούμενους μήνες ε, χάσαμε αρκετό καιρό. Το Συμβούλιο έχει ήδη προχωρήσει και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λιγάκι φιλόδοξοι κυρίως όσον αφορά τεχνικής φύσεως ε, προβλήματα, γιατί εκεί ε, κρύβεται και η πρόθεση να μην εγκρίνεται περιεχόμενο ε, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και στο εξωτερικό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να μην περιοριζόμαστε στο να πιστοποιήσουμε μόνο τους 12 μήνες το Συμβούλιο το έχει και αυτό εξετάσει. Θεωρώ ότι για το Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να πει την άποψή του και έτσι το 2017 να καταλήξουμε μαζί με την κατάργηση της ε, περιεγωγής και την έγκριση της φορητότητας ε, στην Ευρώπη. Ε, τα τεχνικά προβλήματα δεν είναι ανυπέρβλητα. Αν είμαστε φιλόδοξοι νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε κίνητρα έτσι ώστε και οι πάροχοι να βιαστούν λιγάκι και να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να αποφεληθούν νωρίτερα από όλες αυτές τις τις δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Έμα δεν είναι εδώ, ο Ντάν την αντικαθιστά. Εγώ αντικαθιστώ την Έμα σήμερα, είναι σκιώδη συγγήτρια. Πρώτα απ' όλα ε, θέλω να σας πω το εξής. Είμαι σε μια περίεργη θέση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστώ την Κομισιόν που υπέβαλε αυτό που κατά την άποψή μου είναι μια καλή πρόταση. Ευχαριστώ επίσης ε, και τους σχελιστές και το ΕΛΚ. Ε, θέλω να σας πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα. Βεβαίως ε, ο διάβολος υπάρχει πάντα στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι υπάρχει η δυνατότητα του opting in Βέβαια είναι δύσκολο το opting, ε, χωρίς άδεια. Αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στον, ε, στη νομοθεσία. Και επίσης πιστεύω ότι η επαλήτευση είναι το κλειδί για όλο αυτό το θέμα. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με όλα τα σχόλια που έγιναν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει χρονικό όριο, γιατί αυτό αυτό υπονομεύει την πρόταση. Δηλαδή, αν κανείς επιτρέπει τη φορητότητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε κατ' ουσίαν δεν την επιτρέπει. Άρα δηλαδή θα πρέπει να είναι σωστή η επαλήτευση. Και όσον αφορά την ανάγκη για καμία επαλήτευση για το 16, νομίζω πρέπει να ε, πιστούμε πάρα πολύ παν ότι η φορητότητα δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ε, νέες διαπραγματεύσεις για τα συμβόλαια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η επαλήτευση μπορεί να γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποια αντίφαση και ίσω να καθυστερήσει και η θέση σε ισχύ τη πρόταση κάτι που πολλοί από εμά δεν επιθυμούμε. Επίση, ε, αυτό που ε, μα ενδιαφέρει είναι και αν υπάρχει επαλήθευση με default, ε, αν δεν αποδειχτεί ε, το θέμα της ε, μόνιμης κατοικίας, ε, τα πράγματα αλλάζουν ουσιαστικά. Είναι θέμα κλειδί αυτό και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρόταση για να βάλουμε διάφορα παρατηράκια στην πρόταση. Τώρα, οι πάροχοι βεβαίως και έχουν δυνατότητα να καταλήξουν σε μια εναλλακτική συμφωνία στο κρίκετ υπάρχουν πανευρωπαϊκές άδειε, παρότι αυτό δεν παίζεται στην Ευρώπη ε, και ελπίζω ε, αυτά όλα να αλλάξουν. Επίσης, μουσική το, και διάφοροι άλλοι χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι φορητότητα, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τρόπο και αυτό είναι σημαντικό τα πράγματα να ε, βελτιωθούν στην φορητότητα. Δεν πρόκειται για πανευρωπαϊκές άδειες, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, να μην τα μπερδεύουμε. Επίσης, το 8 ε, μας ανησυχεί λιγάκι Νομίζω ότι ενώ είμαστε υπέρ του ε, να υπάρχει η επαλήθευση, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν ε, δυσχεραίνουμε τη δουλειά των εταιριών για να βρουν ε, καταναλωτές. Επίσης, το θέμα των κατεξοδότησης πράξεων, όσο έχουν τα πράγματα τώρα, υπάρχει ο κατάλογος 3β και στο μέλλον ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην πρέπει να παρεμβαίνει. Άρα δηλαδή δεν βλέπουμε ακόμα την ανάγκη ε, να τεθεί το θέμα των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων. Ε, πάντως Αυτά είναι κάποιες από τις ανησυχίες μας, με λεπτομέρειες βέβαια, σε γενικές γραμμές στηρίζουμε τον εισηγητή και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι τελικά ε, θα επιτευχθεί μια καλή συμφωνία. Ευχαριστώ. Thank you. And... Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους τώρα. Η κυρία Τσάνσεβα είναι η συγκήτρια, αλλά καλύφθηκε την κυρία Κάλλας. Την αντικαθιστά η κυρία Κάλλας. Μας μπερδεύουν συνέχεια τη μία με την άλλη. Και μπορούμε να αντικαθιστούμε μία την άλλη να διαβάσω τα δικά της σχόλια. Uh, και μερικά δικά μου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Εξακολουθεί να έχει όμως κάποιες ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα στη γνωμοδίτηση και σε κάποιες άλλες επιτροπές κάποιοι έχουν συμπεριλάβει κάποιες πολιτικές δηλώσεις σε τελογικές σκέψεις, κυρίως για την εδαφικότητα και τη σχετική αρχή. Η ομάδα μου δεν υποστηρίζεται τέτοιες δηλώσεις, όπως στην τροπολογία 2. Για το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλοί στο Κοινοβούλιο αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το κείμενο του Συμβουλίου αντί το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό χρησιμοποίησαν σε βάση για τροπολογίες. Δέχομαι την προσέγγιση, διότι θα επιταχύνει τους μελλοντικού ε, τριμερείς διαλόγους. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία στην εκδοχή του Συμβουλίου που πόρα απέχουν την τελειότητα και λείπουν και στοιχεία. Για χρονικούς λόγους θα εστιαστώ επί του πιο σημαντικού ζητήματος. Δηλαδή ο κατάλογος για την επαλήθευση, ή εξακρίβωση του κρατους μερους μέλους διαμονής. άνθρωπο άρθρο 3β. Και για το κείμενο του Συμβουλίου και στις τροπολογίες της Του συγγητή. Δεν μου αρέσει να έχουμε κατάλογο. Όμως, αν πρέπει να έχουμε κατάλογο, θα πρέπει τα μέτρα να είναι τα λιγότερο δυνατόν δυσδυτικά για να διαπιστώνεται ο τόπος διαμονής. Άπαξ. Από τη στιγμή που ο συνδρομητής έχει εξακριβωθεί ότι μένει εκεί που έχει δηλώσει, όλα είναι εντάξει. Θα πρέπει ίσως να γίνεται έλεγχος διευθύνσεως IP, τη στιγμή συνδρομής ή πρώτης εξακρίβωσης. Αλλά η πρώτη εξακριβωσης αλλα η ομαδα μου δεν θα υπερψηφίσει το μέτρο ως προβλέπεται. Μετά πρόσβαση πρέπει να περιορίζεται στον... Ε, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι στα χέρια του παρόχου αυτού καθεαυτού και, σε όχι, και όχι σε τρίτα μέρη ούτε σε κατόχους δικαιωμάτων. Ούτε αυτοί θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να δουν τα στοιχεία. Τώρα επιλογή επαλήθευσης και τα μέσα επαλήθευσης αυτά είναι στα χέρια του παρόχου υπηρεσιών. Παράγραφος 3 του κειμένου του Συμβουλίου ε, είναι απαράδεκτη. Κάθε παρόχος υπηρεσιών έχει χιλιάδες ε, συμβόλαια με διάφορους κατόχους δικαιωμάτων εφιάλτης για τους παρόχους και για τους συνδρομητές αν κάθε κάτοχος δικαιώματος θα πρέπει να έρθει σε επαφή, μαζί με το, σε επαφή με το συνδρομητή για να επαληθεύσει κατά πόσο προστατεύεται παρκώς και να κάνει επαλήθευση. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά πρέπει να καλυφθούν, θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες, η ΔΙΤΕ θα υποβάλει τροπολογίες. Θεωρεί ότι ο κανονισμός δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τον άλλο κανονισμό για τα πνευματικά δικαιώματα. Η φορητότητα δεν θα πρέπει να φέρει σε δυσχερή οικονομική θέση κανέναν. Δεν θέλουμε να είναι κάτι επιβλαβές για τη δημιουργικότητα στην Ευρώπη και το περιεχόμενο. Θέλουμε απλώς να ευκολύνουμε τη ζωή του απλού πολίτη. Η αντίδραση στι τεχνολογικέ αλλαγέ από τη βιομηχανία ή του πολιτικού δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα μέσα. Αν δεχθούμε το κείμενο του Συμβουλίου θα έχουμε δυσανάλογα μέτρα για να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα για την επαλήθευση θέλω να πω τα δικά μου. Πολλά ήδη υπόθεκαν για την επαλήθευση. Πρέπει να έχουμε υπόψη και κάτι άλλο. Έχουμε ένα κανονικό που είναι και μελλοντοστρεφής. Εάν έχουμε στον κατάλογο κάτι που απαιτεί σάρωση εγγράφων και αποστολή αυτών δεν είναι κάτι μελλοντοστραφές. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας λοιπόν ότι χρειάζονται κατάλληλα μέτρα. Πολλές εταιρείε προβλέπουν δυνατότητα σύναψη συνδρομής στο διαδίκτυο. Θα πρέπει οι εταιρείε να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα ταυτοποίησεως και όχι έγγραφα. Και κάτι άλλο που με ανησυχεί. Η περιοδικός έλεγχος της παροχής των υπηρεσιών μέσω ελέγχου της διευθύνσεως IP ή γεωλογικών στοιχείων, ε, συντεταγμένων μάλλον. Θα πρέπει να ελέγχεται η διεύθυνση ε, IP μόνο μια φορά τη στιγμή σύναψης της συμφωνίας συνδρομής, αλλά όχι κατά την, ε, επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του συμβολέου, τη διάρκεια του συμβολέου. Άλλος, της γούε που θέλει να μιλήσει. Όχι, Γιούλια από τους Πρασίνους. Συγγνώμη, καθυστέρησα βλέπετε. Νομίζω ότι καλά τα πάμε όσον αφορά την πρόταση περιφορητότητας. Είναι σημαντικότατο να διατηρηθεί η αναλογικότητα και να μην δημιουργήσουμε κανόνες που να είναι περίπλοκοι είτε για τους καταναλωτές ή να είναι κάτι επαχθές για τις επιχειρήσεις και τις και να δημιουργήσουμε και άλλο βάρος ε, και δυσχέρεια χρήσεως ε, από τους ενδιαφερομένους. Ενώ αυτό που θέλουμε να κάνουμε την πρώτη φορητότητα είναι να διευκολύνουμε τα πάντα. Να είναι πιο ελκυστικές οι προσφορές για τους καταναλωτές όσον αφορά τις νόμιμες αυτές υπηρεσίες. Καλή αρχή αυτή, δηλαδή να καθορίσουμε χρονικό όριο για τη διάρκεια της φορητότητας, ότι αυτό έχει αποσυρθεί πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο είναι όλα ξεκάθαρα. Δηλαδή ότι οποιοδήποτε έχει μόνο ένα κράτος συνήθους διαμονής. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι παραδείγματα όπου το που είναι η μόνιμη διαμονή τους δεν είναι ξεκάθαρο. Αν κάποιος πήγαινε έρχεται, Φερρυπίν, εργάζεται σε μια χώρα και μένει όμως άλλη χώρα. Ε, είναι πρόβλημα. Ή να έχει ένα διαμέρισμα, να πληρώνει νίκη, κοινόχρηστα κλπ. σε δύο χώρες και να περνάει σε κάθε μέρος σημαντικό χρονικό διάστημα. Τι γίνεται εκεί. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα ότι κάποιοι άνθρωποι διαμένουν κανονικά σε δύο χώρες. Αυτό δεν ξέρω μπορεί να αντικατοπτεστεί στην πρόταση. Στο κάτω-κάτω πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η πρόταση δεν θα πρέπει να είναι και αλεξίσφαιρη. Δηλαδή, το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί αν κάποιο καταχραστεί τον κανονισμό φορητότητος θα ήταν ότι κάποιο θα πληρώνει για περιεχόμενο το οποίο δεν θα έπρεπε να μπορεί να πληρώσει. Αυτό δεν είναι και κάτι πολύ επικίνδυνο σαν ενδεχόμενο, οπότε θα πρέπει να λειτουργούν οι κανόνες, να είναι ελκυστικοί για τους χρήστες και να μην βάλουμε μέτρα διαφύλαξης που θα επιβαρύνουν όλες τι ιδιαίτερε επιχειρήσει ή να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των ε, χρηστών. Με αυτούς τους γενικούς κανόνες υπόψη θα πρέπει να είμαστε σε θέση να περάσουμε αυτή την πρόταση τάχιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο γίνεται να τηρήσουμε το αρχικό εξάμεινο φάσος ε, εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι Είχαν πει τότε ότι ο κανονισμός φορητότητος θα ετίθεται σε ισχύ μαζί με το τέλος των συμπληρωματικών τελών περιαγωγής. Και τότε θα είναι πιο ελκυστικό να χρησιμοποιούν υπηρεσίες του διαδικτύου καταναλωτές όταν ταξιδεύουν, διότι δεν θα έχουν συμπληρωματικά τέλη να πληρώσουν, δεν υπάρχει περιαγωγή. Έχοντας αυτό υπόψη, εφόσον αυτός ο κανονισμός σχετικά απλός και αν τα κάνουμε όλα σωστά, είναι αρκετά εύκολο εφάρμοστος, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σβάμπ παρακαλώ. Ευχαριστώ. θα μπορούσα να αποσύρω ότι παρέμβαση θα είμαι όμως πολύ σύντομος. Νομίζω ένα δίλημα έχουμε μπροστά μας. Και η κυρία Κάλλας που μίλησε για την ε, ε, future proof και για την συνάδελφο που ανέφερε το αλεξίσφαιρο bullet proof, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πρόταση για την φορητότητα του ε, των πνευματικών δικαιωμάτων ε, δεν θα έπρεπε να τροποποιηθεί εκ βάθρων, αλλά να απλουστευτεί περισσότερο. Μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές απόψεις βέβαια, αλλά αν δεχθεί κανείς την απλούστευση ως πρόταση, τίθεται το ερώτημα πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά ώστε στο τέλος ε, οι νομικές απαιτήσει να υλοποιηθούν που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και το copyright σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συζήτηση για την verification process, την επαλήθευση, φυσικά θα πρέπει στην πραγματικότητα της ζωής των νέων ανθρώπων να τη λάβουμε υπόψη. Αλλά το ερώτημα τίθεται. Με αυτή την πρόταση μπορεί να γίνει αυτό όπως ε, μας το ζητούν, όπως ζητείτε ή μήπως θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση που πραγματικά την έδρα ή την κύρια έδρα του πολίτη θα την ε, ε, εξέταζε ως δυνατότητα. Ομολογώ ότι για μένα και για την, τις δικές μου απόψεις για τη μεταφορε, τις μεταφορές στοιχείων δεν μπορώ να σκεφτώ το πώς θα μπορούσε σε σχέση με, τις, ε, με την έδρα να γνωστοποιείται η, έδρα προς τον πάροχο. Θα είχα δυσκολία όσον αφορά τις, τους λογαριασμούς παρόχου με βάση αυτά να τους ελέγχω. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές πραγματικότητες ε, σήμερα στη ζωή και δεν μπορεί κανείς ε, όλα να τα καλύψει, γι' αυτό τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί πιο αποτελεσματικά να καλυφθεί αυτό. Αλλά δεν έχω μια τελεσίδικη θέση ή άποψη από αυτού ακόμα. Ευχαριστώ. Are there any other speakers on this? Υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν να παρέμβουν, παρακαλώ. So just a couple of comments from me that... Ποια σχόλια από μένα και σε κάποιον βαθμό τρεις, τρία, τρεις τομείς έχουν δοθεί από την Επιτροπή σε σχέση με τη φορητότητα και τα δικαιώματα των καταναλωτών ε, και το ψηφιακό περιεχόμενο και θεωρώ εγώ ότι αυτή θα ήταν η πιο σαφής νομοθεσία σχετικά, αλλά βλέπω και εγώ τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ότι θέλουμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες για τους πολίτες σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ε, μηνυμάτων ή ε, παροχών όταν ταξιδεύουν. Δεν θέλουμε να έχουμε την ανεπιθύμητη επίπτωση να περιοριστεί το περιεχόμενο κατά κάποιο τρόπο ή ε, το πολυσχηδές του, των μηνυμάτων που θα πρέπει να μπορούν να διαβιβάζονται. Αλλά και εδώ πραγματικά πρέπει να μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα, το, τη συνολική εικόνα. Και σύμφωνα με την, σφιγμο, την σφιγμομέτρηση πέρσι, μόνο 4%, 4 των καταναλωτών προσπαθούν να έχουν πρόσβαση από άλλο κράτος μέλος. Πάνω από 50% θεωρούν ότι αυτό δεν θα ήταν σημαντικός παράγοντας για αυτούς για τη συνδρομή και εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να μπορούν να έχουν αυτές τις υπηρεσίες ε, ε, ε, στο σπίτι τους. Αυτό θα πρέπει να δούμε από πλευράς περιεχομένου. Να μην υπάρξουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων στην μητρική τους γλώσσα όπως το χρειάζονται. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν να τα κάνουμε σωστά τα πράγματα αυτό, αυτά και νομίζω αυτό συνοψίζει και την άποψή μου. Ο κύριο Ζούλο παρακαλώ τώρα. Αν η Επιτροπή ίσω θα θέλει να παρέμβει πρώτα. Εντάξει, ο Μάρκο Ζούλο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρώτα, Ευχαριστώ του συναδέλφου για τι ε, χρήσιμε προτάσει του. Δάτων τη ευκαιρία για να κάνω μια διευκρίνηση. Για να διαλύσω κάποια αμφισημία, ίσω που να υπάρχει. Για να καθορίσουμε την εξακρίβωση, την επαλήθευση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εντό του κειμένου να καθορίσουμε κριτήρια. Για να καθορίσουμε μέσω των κριτηρίων τη διαμονή. Όχι τα μέσα εξακρίβως. Τι σημαίνει αυτό. Αν εμείς σαν κριτήριο κάνουμε αναφορά, το χάρη στον εργασμό του τηλεφώνου. Ο εργασμός του τηλεφώνου υπήρχε εδώ και χρόνια και θα υπάρχει και σήμερα και θα υπάρχει και στο μέλλον. Αυτό είναι το κριτήριο μέσο θα είναι διαφορετικό. Πριν από πέντε χρόνια ήταν στο χαρτί, ε, ήταν μέσω email. Σήμερα πιθανότατα θα μπορεί να είναι μέσω μια εφαρμογή να πληρώνει το λογαριασμό στο κινητό. Μην μπαίνοντα τώρα στην ουσία του μέσου επαλήθευση, εξακρίβωση, που μπορεί να ποικίλει τεχνολογικό και να αλλάξει γρήγορα, κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα άριστο συμβιβασμό. Η κατεξισοδότηση πράξη θεωρείται καλό εργαλείο για να έχουμε δυνατότητα ενημέρωση επικαιροποίησεως των κριτηρίων μέσω μιας κοινή διαδικασίας. Και ο τομέας μπορεί να συμμετέχει και οι ενώσεις των καταναλωτών. Κάνοντας αυτές τις διακρίσεις λοιπόν, ε, πιστεύω ότι εκείνος που φοβάται ότι ίσω περιοδικά με κάποια συχνότητα θα πρέπει να ε, αλλάζουμε τον κατάλογο των κριτηρίων, αυτό δεν θα γίνει. Διότι από τη στιγμή που έχουμε καθορίσει με σίγουρο τρόπο τα κριτήρια, μετά χωρίς να πούμε στην ουσία των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση, δεν θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διάφορες προτάσεις που κάνατε. Ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο και μετά θα κάνουμε διακοπή, ένα διάλειμμα. Πάμε στο επόμενο σημείο και μετά θα ξεκινήσουμε το Solvit στις 16 και 30. Έχουμε λίγα λεπτά για να συζητήσουμε. The, um, next item agenda, which is the network. Λοιπόν, η οδηγία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, συζήτηση της πρώτης συμβουλίου. Ο Ανδρέας Σβάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να είμαι σύντομο. Τα δίκτυα και η ασφάλεια για την πληροφορία, IT security με άλλα λόγια. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με αυτό. Έχουμε δει τα πράγματα και ε, τον Μάιο το Συμβούλιο ήδη καθόρισε τη θέση του και έτσι επιβεβαίωσε τον συμβιβασμό που σε πρώτη ανάγνωση και ε, νόμιζα ότι ήταν δεύτερη ανάγνωση, αλλά σε πρώτη ανάγνωση αυτό που συμφωνήσαμε με το Κοινοβούλιο, με πρόταση από την παλαιά κοινοβουλευτική θητεία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Είναι σημαντικό βήμα που στον τομέα τη εσωτερική αγορά για την κυβερνοασφάλεια οδηγεί σε αίσιο πέρα. Κάποια σημαντικά στοιχεία βελτίωση προβλέπει όσον αφορά την κέρια υποδομή την ζωτική υποδομή. Υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις ε, που εκείνες που σε σχέση με την οδηγία για την ομοθεσία στα κράτη-μέλη πρέπει να εξεταστούν για την περίπτωση της πολωνικής ε, εταιρείας LOT, και για την και την, τον πάροχο κινητών υπηρεσιών Α1 στην Αυστρία που πάλι λόγω του ότι hackers είχαν ε, προσβάλει αρκετές, επί αρκετές ώρες το δίκτυό του, είχε δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ε, ο ορισμός ε, της κέρια της ζωτικής υποδομής και σε σχέση με την οδηγία που προβλέπει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποφεύγεται στο μέλλον και σε, σχέση με την TV5 της Γαλλίας ή με παρόμοιες περιπτώσεις όσον αφορά την ε, ε, συμπερίληψη αυτών των περιπτώσεων που μπορεί το κράτος μέλος αναπερίπτωση να καθορίζει αλλά ο ορισμός για την εσωτερική αγορά ε, βελτιώνει τα πράγματα όσον αφορά τις ζωτική, τις ζωτικές υποδομές. Έχουμε αρκετές φορές συζητήσει αυτό το θέμα και με τους σκιώδεις εισηγητές που σε αυτό το σημείο στεναρά εξέθεσαν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους μέσω του ορισμού των Digital Service Providers συνεισφέραμε ώστε αυτό για το οποίο συζητούμε σήμερα για την πλατφόρμα νομοθεσίας απλά και ρεαλιστικά να, να έχει επιληθεί. Α, διαφορετικά από τις ζωτικές υποδομές οι πάροχοι μέσω του World Wide Web βρίσκονται σε ειδική θέση όσον αφορά την εξοικείωσή τους με τα θέματα των hackers και της κυβερνοασφάλειας. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει άμεσα να μπορούν να ενημερώνουν τις αρχές. Και νομίζω καθορίσαμε με τη δουλειά μας αυτά τα πράγματα και μπορέσαμε να αποσαφηνίσουμε ότι οι υπηρεσίες παροχή υπηρεσιών σήμερα είτε με αναλογικό τρόπο είτε ψηφιακό τρόπο θα πρέπει να μπορούν να παρέχονται. Αλλά οι υπηρεσίες εκείνες ε, που ψηφιακά θα πρέπει να μπορούν να ε, διαχέονται, θα πρέπει να εξυπηρετούν την κοινωνία της πληροφορίας. Και η εσωτερική αγορά θα πρέπει να ρυθμίζει για τον αναλογικό τρόπο διαβίβασης και τον ψηφιακό τρόπο διαβίβασης τα πράγματα, ώστε εκείνος ο οποίος θα χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες να οδηγείται στο ίδιο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο άλλων εκθέσεων ιδείας πρωτοβουλίας. Θα χαιρόμουν αύριο αν θα μπορούσαμε με μία ε, ψηφοφορία ε, να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε. Θέλω τους ε, συνεργάτες να τους ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές να τους ευχαριστήσω για την υποστήριξή τους. Νίκολα Ντάντη. παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο ΣΒΑΠ. Είμαστε ικανοποιημένοι διότι το Συμβούλιο επιτέλους επίσημα σε αυτή την οδηγία, τη συζητούμε επί καιρών. Πέρασε και πολλής χρόνος από όταν βρήκαμε το Δεκέμβριο του περασμένου έτους το συμβιβασμό. Πέρασε χρόνος λοιπόν. Είναι ικανοποίηση που φτάσαμε σε αυτό το στάδιο. Ολοκληρώσαμε, συνήψα μάλλον σημαντική συμφωνία επί προτάσεως στρατηγικής σημασίας. Αυτά που διαβάζουμε στον τύπο κάθε μέρα σε εφημερίδες και τα διάφορα άθρα αναφέρονται στην ανάγκη της ασφάλειας στο παγκόσμιο αυτό σύστημα που από αυτό εξαρτάται και ασφάλεια των πολιτών στα πληροφοριακά δίκτυα. Χρειάζεται ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι η προπόθεση για όλα αυτά τα πράγματα που ασχολούμαστε σε αυτή την περίοδο, όπω είναι η ψηφιακή αγορά. Εάν δεν υπάρχει ασφαλές δίκτυο, θα είναι λιγότερο ασφαλές το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν θα αναπτυχθεί το εμπόριο το ηλεκτρονικό επαρκώς, δεν θα αναπτυχθεί α, και η διακυβέρνηση ηλεκτρονική, η διάδοση των πληροφοριών κλπ. Όλα αυτά είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Είναι μια οδηγία λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική. Και τελικά η τελική μας θέση με το Συμβούλιο απέχει πολύ από την αρχική θέση του Κοινοβουλίου. Όμως όπως όλα τα πράγματα το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Βρήκαμε έναν καλό συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός αυτός που είναι καλός θα μας δώσει τη δυνατότητα, θα δώσει τη δυνατότητα να θεσπίσουμε κοινού κανόνες και να έχουμε καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια και τις μυστικές πληροφορίες και την ε, συλλογή πληροφοριών. Προβλέπεται στενή συνεργασία των κρατών, επιχειρησιακή στρατηγική. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς και τα κριτήρια για τον καθορισμό των κρισίμων ε, φορέων όπως και η πάροχοι των ψηφιακών υπηρεσιών. Έχουμε τη δυνατότητα και τον τρόπο στα επόμενα χρόνια να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα που θα εγγυάται ασφάλεια στους πολίτες, στους καταναλωτές και στις ευαίσθητες ε, και τις βασικές μάλλον υπηρεσίες ε, τις οποίες απολαμβάνουν. Στην Ολομέλεια, στην ψηφοφορία ε, χρειάζεται για να πετύχουμε τους χρόνους που θέλουμε να κινηθούμε τάχιστα ε, και να επενδύσουμε προσπάθεια σε αυτό το θέμα που είναι στατική σημασία για την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον Ανδρέα Σφαμπ και όλου και όλου εισηγητές για τη συνεργασία και να ευχαριστήσω και τη γραμματεία και τους βοηθούς διότι δεν ήταν κοινή η δουλειά από πλευράς τεχνικής. Επηρέασε πολύ τις δραστηριότητες της Επιτροπής. Σε ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους συνέδραμαν στην πραγματοποίηση αυτού του έργου. Ε, παρακαλώ Σκιώδης, ε, εκ μέρους του ΙΣΤΙΑ πρόκειται για την ε, κυβερνοασφάλεια που για μένα είναι ένας ε, όλο και μεγαλύτερος κίνδυνος για τις κοινωνίες μας, κυρία, κυρίως όταν πρόκειται για υποδομές όπως είναι ο έλεγχος των αερομεταφορών, τα ενεργειακά δίκτυα ή τα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Αυτό λοιπόν, αυτή η νομοθετική ρυθμίση θα επιτρέψει σε όλους να συστήσουν ομάδες, να συνεργαστούν και θα τους βοηθήσει να ε, συνέρχονται οποτεδήποτε χρειάζεται να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές ή όποτε υπάρχει μια υποδομή ε, διασυνοριακή. Πρόκειται λοιπόν για ιδιαίτερα ευαίσθητες ε, διαπραγματεύσεις ε, για να είμαστε πιο ισχυροί. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε, αλλά θα πρέπει και να σεβόμαστε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στη δική μας την εθνική ασφάλεια. Ε, πρόκειται λοιπόν για ε, δύσκολες αλλά πολύ επιτυχημένες διαπραγματεύσεις και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Σβάμπ και την ομάδα των σκιωδών που δούλεψαν μα πάρα πολύ σκληρά ε, για αυτό το, την τόσο σημαντική νομοθετική ρύθμιση. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε και μετά θα ξεκινήσει η δουλειά. Γιατί όπως σας είπα πρόκειται για μια ένα κρίσιμο τομέα όπου η συνεργασία των εθνικών εμπειρογνωμόνων μπορούν να μας καταστήσουν ασφαλέστερους χωρίς να χάνουμε τις εθνικές μας αρμοδιότητες. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ όλους όσοι δούλεψαν πάνω σε αυτό. Άλλος παρακαλώ ή μήπως είναι κάποιος άλλος και όδης ε, εισηγητής παρών. Σας πω ότι ο Τανάς Γιώργα μου ανέθεσε να πω ότι ανεπιφύλακτα υποστηρίζουμε και πολύ θετικά όπως ανέφεραν και συνάδελφοι με θετικό πνεύμα υποστηρίζουμε τη συμφωνία που πέτυχε ο Ανδρέας Σφάμπ επί του θέματος. Μπράβο. Does the Commission wish to say anything? No. Thank you very much. Can we just... Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι ήταν πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις ε, και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει αυτό το αίσιο και έχει έρθει η στιγμή να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας ε, για την πολύ καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο αλλά και με την Προεδρία του Λουξεμβούργου που επέτρεψε να επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα λοιπόν ε, πράγματι πρέπει να περάσουμε στη δουλειά, τα κρατημέλη, για να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η οδηγία. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Πολύ ωραία λοιπόν, θα ψηφίσουμε αύριο και τώρα διάλειμμα για ένα τέταρτο γιατί είμαστε πολύ μπροστά, θα έρθουν οι ε, εμπειρογνώμες κομισιών για να μιλήσουν για το Solvit, θα ξεκινήσουμε στις και μισή. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschusssitzung geht weiter. Leider hat die Vorsitzende gerade einen dringenden λοιπόν, και για την ημερομηνία και γι' αυτό με πα... είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις και με παρακάλεσε εγώ να εκπροσωπήσω, να αναλάβω την Προεδρία και θα το κάνω ευχαρίστω. Ελπίζω να με συγχωρέσουν που στα γερμανικά ομιλώ, στα, στη μητρική μου γλώσσα έχουμε φτάσει στο σημείο, στο scrutiny time της ημερήσιας διάταξης και έχουμε ως θέμα το solve it. Έχουμε προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδιος ως, είναι η Laurence Richemont. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την εισαγωγή, εσάς κυρία Richemont, εισαγωγικά να μας δώσετε τις πληροφορίες εκείνες Πράγμα που γραπτά μας έχετε γνωστοποιήσει και μετά θα παρέμβουν οι συνάδελφοι. Κυρία Αντεορισμού έχετε τον λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Με ιδιαίτερη χαρά προσέχομαι σε εσά για να κάνω αυτή την παρουσίαση για το Europe Advisor και It. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη για το ότι από πλευράς διευθυντού από την Γενική μας Διεύθυνση που θα ήθελε να παραστεί για να παρουσιάσει η ίδια αυτό το θέμα λυπάται που δεν θα μπορέσει να το πράξει σήμερα η ίδια πρέπει να απουσιάσει. Έκανε μια παρουσίαση για την ε, εσωτερική αγορά κάποιους μήνες πριν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο 2015 και μετά από αυτή την παρουσίαση με ένα πιο σύντομο βίντεο για την εσωτερική αγορά και για το Europe Advice και τώρα έχουμε αυτό το βίντεο το οποίο έχει διανεμηθεί στα μέλη της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής και τα καλά μαντάτα είναι ότι ελπίζουμε ότι και στις 24 επίσημες γλώσσες ε, σχετικά σύντομα θα υπάρξει ένα τέτοιο βίντεο ώστε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η ευαισθητοποίηση για αυτά τα θέματα. Τώρα αυτό που θα ήθελα να υπενθυμίσω είναι ότι με τα μέσα και εργαλεία για την εσωτερική αγορά επικεντρωνόμαστε στο να μπορέσει να λειτουργήσει στην πρακτική της συνιστώσας, στην καθημερινή της πρακτική η εσωτερική αγορά. Και από πλευράς Επιτρόπου όταν προσφόρησε την Ολομέλεια τον προηγούμενο Μάιο για την ε, στρατηγική για την ενιαία αγορά επικεντρωνόμαστε στα πραγματικά προβλήματα της πραγματικής ζωής και στοχεύουμε, είναι στοχοθετημένες οι πρωτοβουλίες μας για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και προσκόμματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια πρώτα για το Europe Advice. Τα καλά μαντάτα είναι ότι έχουμε την 20η επέτειο αυτής της πρωτοβουλίας εφέτος και από τη δημιουργία αυτής της πρωτοβουλίας το 1996 πάνω από 200.000 ερωτήσεις υποβλήθηκαν από πολίτες και επιχειρήσεις, οι περισσότερες ήταν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφορούν αυτές οι ερωτήσεις ε, θέματα που απορρέουν από την νομοθεσία και το νομικό πλαίσιο. Και ουσιαστικά έχουμε και πραγματογνώμονες ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άτομα που όταν υποβάλλεται ερώτηση, το πολύ πολύ σε μια εβδομάδα υποβάλλεται η απάντηση σε τέσσερις εργάσιμες μέρες. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία αυτή που και στις 24 επίσημες γλώσσες παρέχεται. Τα πιο συχνά ερωτήματα είναι, για παράδειγμα, τα θέματα τα συνταξιοδοτικά, τα ωφέλη όσον αφορά τον επαγγελματικό βίο, θέματα ασφαλιστικά, θέματα που αφορούν την επαγγελματική ζωή, ε, αναγνώριση διπλωμάτων, πτυχίων όσον αφορά τους εργαζόμενους, ε, οχήματα, καταχώρησή τους κτλ. Πέρυσι το 2015 από πλευράς Europe Advice απαντήσαμε σε 22.000 ερωτήματα που θα έλεγα ότι είναι μια σταθερή αύξηση αυτή και οι απαντήσεις αυτές κομμένες και ραμμένες με, με εύληπτο τρόπο και με εύληπτη γλώσσα καθιστούν την υπηρεσία αυτή μία, ας το πω έτσι με ανθρώπινο πρόσωπο, ερμηνεία του δικαίου και του νόμου. Έχουμε φτάσει στις 200.000 τώρα απαντήσεις. Είναι ένας μεγάλος πλούτος πληροφοριών για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη η νομοθεσία, τα κενά και χάσματα που υπάρχουν για τις προσδοκίες των πολιτών κτλ. Οι πληροφορίες και οι τράπεζες δεδομένων που είναι διαθέσιμες και στην αρχική ή μητρική γλώσσα και στα αγγλικά για την ε, εξέλιξη αυτών των πολιτικών αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τρόπους ε, για την πιο συχνή και πιο ε, ε, αποτελεσματική χρήση αυτών των δεδομένων, των τραπεζών δεδομένων. Δύο λόγια για το Solvit. Solvit, ένα άτυπο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων για πολίτες και επιχειρήσεις όταν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή νομοθεσίας μεταξύ για παράδειγμα δύο κρατών μελών ή κρατικών αρχών. Το Solvit είναι ένα δίκτυο επίσης και βασίζεται σε εθνικά κέντρα Solvit που ε, λειτουργούν στις ε, κρατικές αρχές και υπηρεσίες των κρατών μελών ώστε να βοηθηθούν άτομα και πολίτες ώστε να κάνουν τη βέλτιστη χρήση των δικαιωμάτων τους στην εσωτερική αγορά και να την χάνουν της αρρωγής να αντιμετωπιστούν διασυνοριακά προβλήματα επίσης. Για όλους αυτούς τους λόγους συνεισφέρει πιστεύω σε μια θετική απήχηση και αντιμετώπιση από τους πολίτες για τη διασφάλιση της σωστής ε, μεθόδου και εφαρμογής από τα κράτη-μέλη. Είναι ένα ισχυρό μέσο εν μεταξύ για να μπορεί να λειτουργεί τόπου η εσωτερική αγορά και αυτός είναι ένας λόγος για τους οποίους οι στοχοθετημένες στρατηγικές για την εσωτερική αγορά θα ε, έγκυνται στο να ενισχυθεί το Solvit και αυτό αποτελεί τμήμα της, ε, του ευφυούς πυλώνα εφαρμογής αυτής της στρατηγικής. Και όσον αφορά τα συμπεράσματα ε, του Φεβρουαρίου, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κατεπηγόντως μέτρα και δράση για την ενδυνάμωση, ενίσχυση του σόλβιτ και υπό το φως του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την εσωτερική αγορά και τη στρατηγική της εσωτερικής στην εργασία στο έργο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί, θα προσπαθήσει να ε, ταυτοποιήσει ποιες δράσεις πρέπει να αναλυθούν ώστε να ενδυναμωθεί το Solvit. Μια από τις ιδέες ιδιαίτερα είναι να ταυτοποιήσουμε, να εντοπίσουμε τάσεις ε, στην εσωτερική αγορά και να δώσουμε μια σωστή παρακολούθηση και συνέχεια στα διαθροτικά structural issues, στα διαθροτικά ζητήματα όσον αφορά τον νόμο, την νομολογία και την νομοθεσία, ώστε να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά. Τρεις κύριοι άξονες υπάρχουν όσον αφορά τη δράση για την ενίσχυση. Πρώτον, ενίσχυση του ρόλου αντιμετώπισης παραπώνων, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδυνάμωση, ενίσχυση της συνεργασίας με τα εθνικά κέντρα Solvit που λειτουργούν στα, στις υπηρεσίες των κρατών μελών και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών τρίτων ώστε να, αντιμετω... να μπορέσουμε να έρθουμε στο ύψος του να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών να αναφερθώ σύντομα πώς όλα αυτά λειτουργούν ως μέτρα μέσα του, ε, που λειτουργούν για την εσωτερική αγορά, πληροφορίες, νομική πραγματογνωμοσύνη και συμβουλές ε, για την αντιμετώπιση προβλημάτων και συνεργασία διοικητική. Φυσικά υπάρχει συνεργασία και διασφαλίζει συνεργασία μεταξύ αυτών των εργαλείων και συνεργαζόμαστε με τα ευρωπαϊκά contact centers, κομβικά σημεία επαφής ε, και όπως και για τις περιπτώσεις Solvit μπορούν άμεσα να διαβιβαστούν στη Europe Advice ε, αν χρειάζεται ανάλογα με τις ιδιομορφίες και ανάγκες ώστε να μπορέσουν να διαβιβαστούν εκεί που πρέπει να τύχουν τις σωστότερες αντιμετώπισης. Να τονίσω κάποια ε, σημεία, διότι έχουμε ε, μεγάλο αριθμό και τομεακών δραστηριοτήτων. Έχουμε και ένα φυλάδιο εδώ, it, Success Stories, δηλαδή επιτυχίες ε, όσον αφορά τις επιδόσεις του Solvit. Και το ίδιο και για το Solvit Advice, για τις πρόσφατες περιπτώσεις. Είχαμε έναν Μαλτέζο επιχειρηματία και που ζήτησε νομικές συμβουλές ε, για το τι είδους, τι ύψους ε, ΦΠΑ έπρεπε να καταβληθεί ε, δόθηκε απάντηση για το ποια αντιμετώπιση έπρεπε να δοθεί σε αυτό και αυτό είναι μια ενδυνάμει διευκόλυνση από πλευράς της απάντησης. Enabling answer δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος. Και για το Solvit και έχουμε και παραδείγματα για ε, επαγγελματικές δεξιότητες ή αναγνώριση διπλωμάτων πτυχίων, για παράδειγμα για κάποιον που χρειάστηκε αναγνώριση ε, διπλώματος στην Ιταλία και βοήθεια σε κάποιον Βούλγαρο υπήκο που εργαζόταν στο Λουξεμβούργο ελευθερία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών για την ε, δύο εβδομάδες για παράδειγμα όσον αφορά πορτογαλική περίπτωση ε, για παροχή ε, έργου και υπηρεσίας στη Γαλλία. Αυτά είναι παραδείγματα και κάποια από αυτά εμπεριέχονται σε αυτό το φυλάδιο που σας έδειξα. Ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι για την εσωτερική αγορά έχει καταδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο ώστε να μπορέσει η εσωτερική αγορά να λειτουργήσει αποδοτικά. Και συνεχίζουμε το έργο μας για αυτή τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά. Να αναφέρω επίσης τη διαδικασία, του να, ε, τη διεργασία του να προχωρήσουμε σε μια ενιαία πύλη, ιστοπύλη για την εσωτερική αγορά σε σχέση με τους πολίτες. Παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και συγκεκριμένων ε, ε, στοιχείων ώστε να μπορέσουμε διασυνοριακά να διευκολύνουμε τους πολίτες και στην ψηφιακή εσωτερική αγορά και στην ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εργαζόμαστε ώστε να αστευθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα, ώστε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο υπέρ των πολιτών και να τους διευκολύνει. Με όλα αυτά νομίζω ότι μπορώ να επαρκεστώ και να πω ότι εντάξει αναμένουμε σίγουρα υψηλό βαθμό αποδοχής και υποστήριξης από τους ευρωβουλευτές αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την περαιτέρω μετεξέλιξη και ενίσχυση αυτών των μέσων και εργαλείων. Σας ευχαριστώ εκ προημίου για την υποστήριξή σας και για τη βοήθειά σας. Είμαι σίγουρη ότι κάποια μέλη θα έχουν ερωτήσεις την αρχή δώσατε κάποια στατιστικά στοιχεία. Εγώ περίμενα περισσότερα στατιστικά στοιχεία και μία παρουσίαση από πλευρά σας. Μας παρουσιάσατε λοιπόν την ενημέρωση, την έκθεση, την τριμηνία. Δεν... Υπάρχει μία έκθεση τριμηνία, έτσι δεν είναι. Δεν την παρουσιάσατε αυτή, ναι. Τα βασικά στοιχεία που παρουσίασα στην εισαγωγή μου είναι ότι απαντήσαμε σε Europe Advice σε 200.000 ε, ερωτήσεις. Πέρσι ήταν 22.000 ερωτήσεις. Μπορούμε να δώσουμε λεπτομερέστερα στοιχεία μέσω της τριμηνίας εκθέσεως. Αν πάρουμε το πρώτο τρίμηνο του 2016, από 5.769 υποθέσεις αποδεκτές, που κωδικοποίησαν οι πυρογνώμονε. 740 ενδιαφέρουσες υποθέσεις συμπεριλήφθησαν στην έκθεση, διότι η έκθεση δεν καλύπτει όλα τα θέματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. 6.000 ερωτήσεις απαντήσαμε το πρώτο τρίμηνο. Αναλύονται στις τριμηνίες εκθέσεις σε θεματικές κατηγορίες και γίνεται ανάλυση συνέχεια που δόθηκε στα ερωτήματα αυτά. Αναλύουμε την ταχύτητα των απαντήσεων. Έχουμε σχετικά στοιχεία. Η ερώτησή μου, λέει η Πρόεδρος, οι ερωτήσεις μου μάλλον. καταφθάνουν περισσότερες ερωτήσεις στο Solvit. Πόσες από τις ερωτήσεις που μπαίνουν στο Solvit βρίσκουν λύση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς με προβληματική, διαφορετικοί τομείς προβληματικοί στα διάφορα κράτη-μέλη. Εάν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών. Ξέρω ότι το Solvit βοηθάει πολύ και καμιά φορά όμως δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Υπάρχουν προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη, υπάρχουν προβλήματα σε κάποιους τομείς, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Ίσως άλλοι έχουν ερωτήσεις. Δείτε. Ευχαριστώ. Μπορείτε να βασιστείτε στην ε, στην υποστήριξή μας. Έχουμε και ευθύνε όμως. Θέλουμε αυτά τα εργαλεία, πώς να το πω, να είναι φιλικά. Μ' ακούτε? Έλεγα να είναι φιλικά, προσβάσιμα. Αυτό ήταν το περσινό μου σχόλιο. Όταν επεσκέφθην την ιστοσελίδα σας δεν ήταν ξεκάθαρο πώς γινόταν διασυνδέσεις με κάποιες ε, υπηρεσίες μέσω των links. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Πώς μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο φιλικό προς το χρήστη το σύστημα. Ωραία. Έχουμε τα εργαλεία, τα ξέρετε, τα ξέρουμε. Όμως τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, ώστε να είναι πιο ορατά στο ευρύτερο κενό τα εργαλεία. Αν μιλάτε με αυτούς που ζουν στη Φυσαλίδα, στην Πομφόλιγα των Βρυξελών, ε, τα γνωρίζουν. Αλλά έξω από αυτό τι γίνεται. Μπορούμε να το αναθέσουμε στα κάτι μέλη, όχι. Μπορούμε να προωθήσουμε το εργαλείο αυτό, να το μάθουν οι πολίτες, να ξέρουν ότι υπάρχουν τα εργαλεία. Τι κάνατε στον τελευταίο αυτό χρόνο για να προωθήσετε αυτά τα εργαλεία. Αυτή είναι η ερώτηση. Ε, κυρία Γιακονσάρη, ο άντρας, έχει κάποιες ερωτήσεις. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε σχετικά με το Solvit, νομίζω ότι το ποσοστό επιτυχίας για την απάντηση σε περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί ανέρχεται στο περίπου 80% και για το εναπομένον 20% αυτές είναι κυρίως οι περιπτώσεις που ανέφερα, δηλαδή όπου υπάρχουν ε, διαρθρωτικής ε, φύσης ε, θέματα, παραβίαση ενός νόμου, θέματα που πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Και το θέμα είναι ότι στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί το Solvit, η Κομισιόν προσπαθεί να επιλύσει αυτά τα θέματα που δεν έχουν επιληθεί με το Solvit και το κάνει αυτό εξετάζοντας ε, όλες ε, τις ε, δυνατότητες που υπάρχουν για συνέχεια και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Άρα υπάρχει διάλογος ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κέντρα Solvit για να διαπιστωθεί τι μπορεί να γίνει περαιτέρω σε επίπεδο κρατών μελών. Ίσως για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ή αν χρειάζεται να προσαρμοστεί η νομοθεσία και υπάρχει και ε, διάλογος με όλες τις σημαντικές υπηρεσίες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ε, για να αντιμετωπίσουμε διαρθρωτικής φύσεως θέματα. Όσον αφορά τώρα στο ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να γίνουν πιο φιλικά και πιο προσιτά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και για το ότι αντιμετωπίζετε το θέμα του συσχετισμού ανάμεσα στις ε, διάφορες υπηρεσίες. Μάλιστα, εμείς δουλεύουμε πάνω σε μια προσέγγιση cascade, όπως λέγεται, δηλαδή οι υπηρεσίες συνδέονται πρώτα με το Europortal και αν δεν βρουν απάντηση στο Europortal ε, που είναι βασικές προφορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε όλα αυτά μπορούν να αναδιοχετευτούν στο Europe Advice. Και εάν το όλο θέμα είναι πιο περίπλοκο και ε, προϋποθέτει και άλλα κράτη-μέλη, ε, τότε όλο αυτό καταλήγει τελικά στη Solvit. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε ακόμα πιο εξορθολογισμένα και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι υπηρεσίες ε, περνάνε μέσα από το Europe First και αν χρειαστεί μετά ε, αναδιοχετεύονται σε άλλες υπηρεσίες. Γιατί το θέμα είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ε, κάποια ερωτήματα <clears throat> τα οποία μπορούν να επιληθούν Άρα δηλαδή εμείς ε, προσπαθούμε αυτή τη διασύνδεση να την καταστήσουμε ε, πιο αποτελεσματική και φιλική προς το χρήστη ε, για τις υπηρεσίες και για τους πολίτες. Όσον αφορά το κατά πόσο είναι ορατά όλα αυτά τα εργαλεία στο ευρύτερο κοινό, να σας πω ότι έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για να προωθούν αυτά τα εργαλεία. Υπάρχει αυτό που αποκαλούμε νέοι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας, κυρίως ε, μέσα από την αλλαγή της ε, βελτιστοποίησης του Europortal. Ε, και πρέπει να σας πω ότι επενδύουμε αρκετά για τη βελτιστοποίηση που σημαίνει ότι όταν ο πολίτης έχει μια ερώτηση μπορεί την ερώτησή του αυτή να την βάλει μέσα στο Google ή σε άλλο δίκτυο και να ε, αναδιοχετευτεί στο Europortal. Δεχόμαστε πολλές τέτοιες αιτήσει. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά αποτελεσματικό γιατί βλέπουμε ουσιαστική αύξηση των χτυπημάτων στο Europortal. Έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο χτυπήματα το μήνα, άρα 12 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυξάνεται συνεχώς αυτός ο αριθμός των χτυπημάτων. Βελτιώνεται λοιπόν η βελτιστοποίηση. Κάνουμε πολλά και με το Facebook και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Twitter και ούτω καθεξής. Πρόσφατα οργανώσαμε ένα chat για επαγγελματικά προσόντα και αυτό έγινε ε, σε συνδυασμό με πυρογνώμονες από το Europortal και το Europe Advice. Πολύ επιτυχημένο αυτό το chat ε, πρέπει να σας πω. Είχαμε πάνω από 2.000 ενεργούς μετέχοντες σε αυτό το chat και αν δείτε τα στοιχεία ήταν, είναι ακόμα περισσότεροι, άρα μεγάλη επιτυχία. Αυτά είναι παραδείγματα του πώς προσπαθούμε να καταστήσουμε τα εργαλεία πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ε, σε πολίτες και επιχειρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν ε, διαφορετικά ακροατήρια, υπάρχουν διάφοροι στόχοι. Υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο κατά την άποψή μου ε, το ακροατήριο αυτό είναι οργανώσεις σε κρατημέλη που ενδιαφέρονται ε, ενδιαφέρονται για ε, συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση μέσα από επαφές, ε, παρουσίες. Υπάρχει βέβαια και το ευρύτερο κοινό και γι' αυτό το κοινό πιστεύουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνεται ουσιαστική χρήση όλων αυτών των εργαλείων. Σας ευχαριστώ πολύ. I was looking at your, um, Τι γίνεται με τα διάφορα εργαλεία στις ε, χώρες μέλη και όχι μόνο για το Solvit. Διερωτώ ε, κατά πόσον έχει εντοπιστεί το κόκκινο σε κάποια περιοχή, σε κάποια χώρα και αν εντοπιστεί αυτό, τι γίνεται ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι ορισμένες περιοχές ε, παραμένουν δυστυχώς ε, κόκκινες. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε για να ασκήσουμε πίεση σε αυτό. Κυρία Πρόεδρε, Πράγματι, ε, πάντα μπορεί να υπάρξει πρόοδος από πλευράς κρατών μελών. Εμείς ε, ελέγχουμε όλα τα εργαλεία της ε, ενίας αγοράς μέσα από το βαθμολόγιο. Υπάρχει ένα γράφημα με τα χρώματα του κώδικα κυκλοφορίας όσες χώρες έχουν κόκκινο δεν έχουν κάνει τίποτα και όσοι έχουν πράσινο έχουν κάνει πάρα πολλά. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά τέτοια εργαλεία και πιστεύουμε ότι όλα αυτά βοηθούν έτσι ώστε να σκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη. Γιατί όταν δημοσιεύεται το βαθμολόγιο και το φετινό θα ε, δημοσιευτεί αρκετά νωρίς, ε, τώρα βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης με την Κομισιόν, όταν λοιπόν θα έχουμε την τελική συμφωνία θα δημοσιευτεί. και όταν δημοσιευτεί ε, στα κρατημέλη θα σκηθεί ένα είδος ε, πίεσης Βεβαίως εμείς ε, παρακολουθούμε το διάλογο σε όλες τις συναντήσεις που έχουμε με εκπροσώπους των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει ε, κανονικές συναντήσεις, το Σόλβι συναντιέται δύο φορές το χρόνο με εργαστήρια σε όλα τα κράτη-μέλη μια φορά το χρόνο στις Βρυξέλλες και την δεύτερη φορά σε κάποιο κράτος μέλος. Και εκεί προσφέρει τη δυνατότητα να εξετάσουμε όλα τα θέματα. Αν είναι λοιπόν σημαντικά τα θέματα, ε, μπορούν να εξεταστούν. Επίσης για το Europe Advice Network έχουμε συναντήσεις με αυτό το δίκτυο και αυτό επιτρέπει τη δυνατότητα να κάνουμε training και να εντοπίσουμε και κάποιες μελλοντικές δυσκολίες. Άρα δηλαδή μέσα από την πίεση που ασκούμε ε, μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Και βεβαίως θα ήμασταν πάρα πολύ ευτυχείς να συνεργαστούμε με αυτή την Επιτροπή για να ε, βελτιωθεί περισσότερο η κατάσταση με τα κράτη-μέλη. Μήπως ε, να μας ε, να πείτε στην γραμματεία της Επιτροπής το πώς καταφέρνετε να ασκήσετε πίεση στα κράτη-μέλη γιατί ε, εφόσον θα υπάρχει η νέα έκθεση του δημοσιευτεί και τα νέα χρώματα, το νέο χρωματολόγιο, ε, θα πρέπει να πείτε σε κάθε μέλος του Κοινοβουλίου τι ακριβώς κάνει το κράτος του για να έχουμε μία σαφή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας. Γιατί ε, καλά τα κάνουμε ε, όταν ε, ελέγχουμε την κυβέρνηση, κυρίως όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά θα πρέπει να ε, ξέρουμε και τι κάνουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Γραμματεία της Επιτροπής για να οργανώνουμε συναντήσεις με ευρωβουλευτές που ενδιαφέρονται για να εξετάσουν το θέμα και για να ασκήσουν πίεση στο κράτος τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά για σήμερα. Τελειώσαμε. Αύριο ξεκινάμε στις 9.30. Γεια σας.